Η Πρόεδρος, καλό σας απόγευμα σε όλους και όλους. Σας αρχίσουμε αμέσως την έκτακτη συνεδρίαση. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που έχουμε την ευκαιρία αυτή και που έρχεστε όλοι εσείς να συμμετάσχετε. Να... Ανακοινώσω μόνο ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν βουλγαρικά. Δεν ε, μπορείτε να ακούτε τα βουλγαρικά. Όμως ακούτε όλες τις άλλες γλώσσες. Χαίρομαι πολύ σήμερα που έχουμε κοντά μας τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Τίμερμανς, και μάλιστα για τέταρτη φορά, μέσα στα πλαίσια του διαθρωμένου διαλόγου, ο σκοπός, ως γνωρίζετε, είναι να προβούμε σε μια καταγραφή της προόδου που έχουμε επιτύχει ως τώρα σε ορισμένα θέματα κλειδιά, για τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων γενικότερα και βέβαια να δούμε, να πούμε και λίγα λόγια για το τι αναμένουμε ακόμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βεβαίως και τι αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από εμάς. Και ίσως μπορούμε να πούμε και λίγα λόγια για την επικείμενη, ε, για την επόμενη δηλαδή θητεία. Λίγα λόγια σχετικά με τη διαδικασία. Μετά από το σημερινό διάλογο θα συντάξει η Επιτροπή μας ορισμένα βασικά μηνύματα τα οποία θα διαβιβαστούν στην Πρόεδρο και στην Γραμματεία για την συνοπτική έκθεση για το 2018 και αυτά θα κυρωθούν από την ΙΣΙΣΥ και μετά θα προχωρήσουν στη διάσκεψη Προέδρων Πολιτικών Ομάδων. Έχοντα διευκρινίσει τα πράγματα αυτά, πολύ ευχαρίστω να σα δώσω το μικρόφωνο, κύριε Αντιπρόεδρε, για να προχωρήσετε σε μια εισαγωγική τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με δέχεστε και πάλι βρίσκω την ιδέα καλή, ε, την ιδέα της ανταλλαγής απόψεων, της ε, καταγραφής, της πρόοδου και πιστεύω επίσης ότι εάν αναλύσουμε τις αναφορές που λαμβάνετε και εσείς και ε, μας διαβάζετε και μας, βλέπουμε και πολύ feedback σχετικά με τα αποτελέσματα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σχετικά με τις προσδοκίες που έχουν πολλοί πολίτες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά φορά οι προσδοκίες αυτές είναι τεράστιες και υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητές μας. Το γεγονός όμως ότι απευθύνονται σε εμά, αναφέρονται σε εμά, στους θεσμούς μας, δείχνει ότι έχουν υψηλές προσδοκίες από την δράση μας και ελπίζουν ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί εξ αυτών. Και οι προκλήσεις αυτές απηχούνται άλλωστε συχνά στις αναφορές και στις άλλες επαφές που έχουμε με τους πολίτες μας. Είναι δύσκολη καιρή, πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλοί άνθρωποι ανησυχούν ποια θα είναι η θέση τους στον αυριανό κόσμο και τι μορφή θα λάβει το μέλλον, αν θα έχουν δουλειά τα παιδιά τους. Πρόκειται για υπαρξιακά σχεδόν ερωτήματα που θέτουν τόσοι πολλοί πολίτες και καθημερινά. Είναι, απηχούνται μάλιστα και στη διαδικασία του διαλόγου που έχουμε ξεκινήσει στη βάση της Λευκής Βίβλου ε, έχουμε καταθέσει έναν αριθμό σεναρίων που μπορούν να σκεφτούν όσοι επιθυμούν και να καταθέσουν και τα δικά τους άλλωστε και στη χθεσινή ημέρα που ε, καταθέσαμε το σχέδιο για το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο και όπου βλέπετε και πάλι ότι ε, από την οπτική σας θέση διαμορφώνεται και η γνώμη σας. Αν είστε καθαρός συνεισφορέας και αντιμετωπίζετε τις συνέπειες ε, του Brexit που θα αφήσει ένα μεγάλο κενό στον κοινοτικό προϋπολογισμό, ως καθαρός συνεισφορέας λέτε ναι μεν, αλλά δεν θέλω να πληρώσω περισσότερο. Αν είστε δικαιούχος, ε, λέτε ναι, το βλέπουμε το κενό, αλλά δεν θέλουμε να πάρουμε λιγότερα. Και τα μέλη λοιπόν του Συμβουλίου και της, ε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λένε θέλουμε ισχυρότερε πολιτικέ για την ασφάλεια, για τη μετανάστευση. Αλλά χρειαζόμαστε και τι παλιέ πολιτικέ. Άρα προσθέτουμε όλο και περισσότερε προτεραιότητε και ορισμένε φορέ δεν είμαστε στη θέση να αλλάξουμε τι προτεραιότητε ορισμένων πολιτικών. Αν τα βάλει κανεί όλα αυτά λοιπόν, καταλήγει να είναι ασύμβατα και με την φύση της ευρωπαϊκής Ενωποίησης, η οποία δεν γίνεται βεβαίως με επαναστατικά βήματα, αλλά με εξελιχτικά βήματα και με αναζήτηση συμβασμών. Και αυτή θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε τα επόμενα λίγα χρόνια. Και γι' αυτό είναι σαφές για μένα ότι τα όσα προτείνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρκούν όσον αφορά τον συνολικό προπολογισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως είναι όμως από την άλλη μεριά υπερβολικά πολλά για ορισμένε χώρε μέλη και μάλιστα και τη δική μου τη χώρα και καμιά φορά ο κόσμο εύχεται να έχει νέε πολιτικέ και τι χρειαζόμαστε πραγματικά εν ώψη των προκλήσεων. Άλλοι θέλουν να διατηρηθούν τα πράγματα ακριβώ όπω είναι για να προστατεύσουν τα κεκτημένα Του. Βρισκόμαστε σε μια ήπειρο όπου πολλοί ακόμη αναμένουν να κερδίσουν αλλά και πολλοί φοβούνται ότι θα χάσουν και μέχρι και τα πάντα. Και γι' αυτό οι άνθρωποι προσπαθούν να προστατεύσουν τα κεκτημένα και είναι λιγότερο διατεθειμένοι να μοιραστούν με άλλου. Και μέσα στα πλαίσια αυτά, νομίζω, οι αναφορέ είναι η άμεση οδός επικοινωνίας με τους πολίτες μας και επομένως πολύ σημαντική. Νομίζω ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι οι ανησυχίες που θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να τους προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους βοηθήσει να προοδεύσουν, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε με βελτιωμένη νομοθεσία στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, περισσότερη διαφάνεια, καλύτερη εφαρμοσιμότητα, να αποφευθούν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις και γι' αυτά λαμβάνουμε πολλές αναφορές. Είχα και μια task force φτιάξει, όπως γνωρίζετε, να εξετάζει θέματα επικουρικότητας και αναλογικότητας. Και οφείλω να πω εδώ και πάλι ότι δυστυχώς το γεγονός αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην task force. Και επαναλαμβάνω ότι έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Αν αλλάξετε πολύ ευχαρίστω, αν αλλάξετε γνώμη δηλαδή, πολύ ευχαρίστω να προσέλθετε και να συμμετάσχετε. Τα Εθνικά Κοινοβουλία συμμετέχουν ενεργά, το ίδιο η Επιτροπή Περιφερειών και αναζητούμε τρόπους να εξυγχρονίσουμε την επικουρικότητα και αναλογικότητα. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε από εσά μάλιστα συχνά είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Έχουμε καταθέσει πρόταση τώρα εμεί για την βελτίωση τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ευχαρίστω θα ακούσω τι απόψει σα για το πώ μάλλον αν νομίζετε ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, είμαι σε πολύ στενή επαφή με τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί θέλω... Μάλλον ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να μην περιμένω δική σας έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, αλλά να προσπαθήσω να ευθυγραμμίσω την πρότασή μας με τη δική σας ιδέα πρωτοβουλία, γιατί ελπίζω ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος των θητιών μας και της δικής μα και τη δική σα γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να μπορούμε να δείξουμε στο κοινό, στο ευρωπαϊκό κοινό πριν από τις ευρωεκλογέ. Ότι ακούσαμε όλες αυτές τις ε, μη κρατικέ οργανώσεις που ήθελαν να προωθήσουν κάποια πράγματα και αυτή είναι η πρότασή μας. Βλέπω ότι ο κύριος Βαλένσα είναι παρόν, έχει παίξει εξαιρετικά επικοδομητικό, θετικό, ενεργό ρόλο εξ ονοματό σα. άνθρωπος ιδιαίτερα ρεαλιστής, που ε, κάνει μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων και τον ευχαριστώ. Πολύ επαγγελματίας ε, και πολύ υποστηρικτικός και του είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων. Τέλος, λίγα λόγια για τις διαδικασίες για παραβίαση. Γνωρίζω ότι θέλετε να πείτε, να θέλετε μάλλον να πω κάτι σχετικά. Έχετε κατ' επανάληψη ζητήσει να μιλήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει προσπάθειες να δώσει γραπτές απαντήσεις στο Κοινοβούλιο. Οποιαδήποτε διασύνδεση, διασύνδεση πάντως μεταξύ κάποιων αναφορών και των διαδικασιών που κινούνται στη βάση υπόθεσης παραβίασης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και νομίζω ότι έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιώσουμε την διαφάνεια για τις ε, διαδικασίες παραβιάσεων. Το 2014 έχουμε φτιάξει μια, κεντροποιημένη πλατφόρμα στο Europa website. Συνεχίζουμε να δίνουμε και στα κοινοβούλια και στο κοινό σε βάθος πληροφορίες για την παρακολούθηση της εξέλιξης ευρωπαϊκής νομοθεσίας και για το follow-up που δίνεται. Παρών σήμερα εδώ για να ακούσω από εσά πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Συμφωνούμε εξάλλου απολύτω, ότι οι διαδικασίε για παραβίαση πρέπει να αντιμετωπίζουν θέματα ταχύτατα, να διερευνώνται οι ενδεχομένε παραβιάσει τη νομοθεσία. Αυτό έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε με πιο στρατηγικό και συνολικό τρόπο, όπως άλλωστε και στην ανακοίνωσή μας του Δεκεμβρίου 2016 και ελπίζω να έχω την υποστήριξή σας. Τώρα ευχαρίστω θα ακούσω σχόλια και ερωτήσεις και θα σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Οι συνάδελφοί μου πράγματι ενδιαφέρονται πολύ να συνεχίσουν το διάλογο μαζί σας. Θα παρακαλέσω πρώτα οι συντονιστές να λάβουν τον λόγο και αμέσως μετά θα δώσω τη δυνατότητα να λάβουν το μικρόφωνο και τα υπόλοιπα μέλη. Ο Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν είστε η πρώτη φορά στην ε, Επιτροπή μας. Ε, θέλετε να δημιουργηθεί αυτός ο διάλογος. Ε, εμείς χαιρόμαστε πάντα όταν έρχεστε στην Επιτροπή μας και όποτε θέλετε μπορείτε να έρχεστε. Η πόρτα, μας είναι ανοιχτή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η διμερής συνεννόηση που έχουμε. Μιλήσατε πριν για το πού βρίσκονται οι χώρε ε, για τη μελλοντική, το μελλοντικό προγραμματισμό και ότι εξαρτάται η θέση του από το αν είναι δικαιούχοι, αν είναι συνεισφέροντε. Ε, Βεβαίω υπάρχουν και χώρε που θέλουν να δίνουν λίγα, να παίρνουν πολλά. Υπάρχουν κάθε είδου απόψει. Εν πάση περιπτώσει, για τι αναφορέ. Η Επιτροπή Αναφορών είναι όντω ένα δείκτη για το ότι ζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτε στρέφονται σε εμά με το πρόβλημά του και θέλουν βοήθεια. Είναι καλό δηλαδή να υπάρχει η Επιτροπή των Περιφερειών, γιατί πραγματικά μπορούν να αποταθούν σε αυτή οι ε, πολίτες μας. Ε, είναι ένα δείγμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωντανή. Και βεβαίω ε, πρέπει να απαντούμε στι αναφορέ που γίνονται. Έχω γράψει εγώ κάποια σχόλια για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Νομίζω ότι και ο συνάδελφο Βαλέσσα θα πει κάποια πράγματα μετά. Οπότε του το αφήνω γιατί είναι καθήλυνα αρμόδιο. Δεν θέλω να ανακατευτώ στα χωράφια του. Αυτό που θα ήθελα, τέσσερις μικρές επιθυμίες έχω, κύριε Αντιπρόεδρε. Αυτό που θα επιθυμούσα λοιπόν πρώτα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντά πιο γρήγορα στις αναφορές. Ξέρετε ότι πάει η, Επιτροπή, η αναφορά στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν γρήγορες απαντήσεις, ε, που να μην λένε όμως δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, το θέμα τη αρμοδιότητα, ναι, πρέπει να, γίνει, να γίνεται, να διεκπαιρεώνεται γρήγορα. Πολλέ φορέ δεν συμφωνούμε απολύτω μαζί, μας, μαζί σα, αλλά τώρα, αν περιμένουμε και κάποιου μήνε να δοθεί απάντηση, καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Καλό λοιπόν θα είναι να δίνονται απαντήσει πιο γρήγορα. Δεύτερον, μιλήσατε για τι διαδικασίε επί παραβάση και την παραβίαση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, παίρνουμε μία αναφορά, α πούμε, και η Κομισιόν λέει ναι, ναι έχουμε, σημειώσει, έχουμε σημειώσει ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει παραβίαση τη νομοθεσία και ξεκινάει η διαδικασία παραβάση. Αυτό είναι το βασικό, η βασική είδηση. Αλλά μετά δεν ξέρουμε τι ακριβώ κάνετε. Έχουν στραφεί και προ την πρόεδρο ε, οι συνάδελφοι να ζητήσουν και άλλε πληροφορίε. Εμεί δηλαδή μπορούμε να εμπλακούμε σε αυτό το μετέπειτα στην, στη συνέχεια τη διαδικασία. Γιατί πρέπει να ξέρουμε πώ παρακολουθείτε αυτή τη ε, διαδικασία. Χρειαζόμαστε λοιπόν πληροφόρηση για να μπορεί κάποια στιγμή να κλείσει η αναφορά, να λυθεί το πρόβλημα που αποτελεί το αντικείμενο της αναφοράς. Να ξέρουμε ότι έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατόν να κάνουμε. Μετά, παλιό πρόβλημα που μας ε, απασχολεί πολλές φορές και αρκετά συνηθισμένο σε ό,τι αφορά αναφορές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Υπάρχει ένα project περιβαλλοντικό, το οποίο όμως δεν, αντικαθιστά, δεν, ε, δεν συμβαδίζει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μπορούν να διορθωρθούν κάποια πράγματα που είναι λάθος και η Κομισιόν αυτό που λέει πάντα είναι ότι αυτή τη χρονική στιγμή, επειδή βρισκόμαστε στη φάση του σχεδιασμού, δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε ότι το κράτος μέλος τηρεί την νομοθεσία. Και αυτό σωστό είναι. Από θέμα αρχής είναι σωστό. Είναι καλό να το ξεκαθαρίζει αυτό η Κομισιόν στο κράτος μέλος. Από την άλλη όμως, όταν όντω προχωρά το project, και μπορεί να έχει ολοκληρωθεί ας πούμε μετά από τρία χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναθεωρηθεί το οτιδήποτε. Οπότε καλό θα ήταν να υπάρχει μια πιο εντατική συνεννόηση με, την, με το κράτος μέλος στην φάση της, του προγραμματισμού. Για να, για την, για πολύ αργά να αλλάξουμε το οτιδήποτε. Ο, η, η εγχείρηση μπορεί να έχει πετύχει, αλλά τελικά ο ασθενής απέθανε. Οπότε έχετε το και αυτό υπόψη σας, κύριε Αντιπρόεδρε. Και επίσης ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί έχει να κάνει με το δίκτυο που έχουμε δημιουργήσει εδώ στην ε, Επιτροπή, που πραγματικά έκανε πολύ καλή δουλειά η πρόοδος, γιατί είπαμε ότι πρέπει να μπορούμε τη δουλειά μας που περιλαμβάνει πάρα πολλά πρακτικά προβλήματα, να μπορούμε να την κάνουμε από κοινού σε συνεργασία με τις το, ε, επιμέρους αρμόδιες επιτροπές. Οπότε θέλουμε καλύτερη, πιο στενή συνεργασία. Καμιά φορά καταλήγουμε στο αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βοηθήσουμε στην αναφορά. Γιατί δεν συνάδει η αναφορά με την νομοθεσία, αλλά καμιά φορά είναι και το πρόβλημα της νομοθεσίας που δεν μπορεί να βοηθήσει. Οπότε πώς μπορούμε να έχουμε μία δίωδο επικοινωνίας. Αν πρέπει δηλαδή η νομοθεσία να αλλάξει για να βοηθήσουμε να λυθεί το πρόβλημα του ετούντος. Τι κάνουμε. Η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις νομοθεσίας, αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα συναλλαγής και επικοινωνίας. Ε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ξέρω ότι πολλοί θα θέσετε αρκετά παρόμοια θέματα. Αν ωστόσο έχετε, έχετε παρόμοια θέματα να θέσετε, ε, μην, μας, ε, μην τα αναφέρετε. Μιλήστε μόνο για τα διαφορετικά που έχετε να πείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω διάφορα να πω και δεν θα είναι τα ίδια που είπε ο Πίτερ γιατί μάλλον δεν έχουμε τον ίδιο στόχο. Ο στόχος μας δεν είναι να κλείνουμε τις αναφορέ, αλλά να απαντήσουμε στα θεμητά αιτήματα των πολιτών όταν πρόκειται για λάθος εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να αποκαταστήσουμε τη ζημιά που έχουν υποστεί. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπογραμμίσω φιλικά, γιατί όντως έχουμε πολλές προσδοκίες από το δικό σας θεσμό. Θέλουμε κάποια σημεία να σας πούμε για τα οποία θέλουμε περισσότερα. Γιατί μέσω της Επιτροπής Αναφορών είμαστε ένας υποδοχές ε, των προσδοκιών, των εντόνων προσδοκιών των πολιτών, που δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη, ωστόσο, από το σύνολο των θεσμών. Γιατί ακριβώς το Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής Αναφορών λαμβάνει τα αιτήματα αιτήματα αυτά, αλλά αυτά τα αιτήματα απευθύνονται στο σύνολο των θεσμών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εσεί εκπροσωπείτε μέσω τη λειτουργία της, το ρόλο της που προβλέπεται από τι συνθήκες, είναι ο θεματοφύλακα των συνθήκων και εγγυάται την ορθή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Και είναι αλήθεια ότι μία ακρόαση μετά από ακρόαση ε, έχουμε ενώπιόν μας όλο ένα και περισσότερες περιπτώσεις όπου έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιο είδους ε, υποχώρηση ε, από αυτήν την βασική της λειτουργία της Κομισιόν, δηλαδή την εγγύηση της ορθής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Και όλος ιδιαίτερος έχουμε την αίσθηση πως επικρατεί μια ευαρέσκεια ε, στα κράτη-μέλη όσον αφορά την μεταγραφή των δικαιωμάτων των πολιτών. Για παράδειγμα, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι στη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας εδώ στην Επιτροπή μας, οι προθεσμίες εφαρμογής, για παράδειγμα, για την οδηγία για την ποιότητα του αέρα, που είναι από το 2008, έχει ξεπεραστεί, ε, έχουν ξεπεραστεί αυτές οι προθεσμίες ε, χωρίς να έχει υπάρξει καμία σχετική ε, νήξη από πλευρά τη Κομισιόν ή για το συντονισμό των, κοινωνικών, ε, των συστημάτων κοινωνική πρόνοια, η οδηγία για τα, την ελεύθερη κυκλοφορία. Υπάρχουν ένα σωρό παραδείγματα και είναι αλήθεια ότι θα θέλαμε πραγματικά να υπάρξει ίσως μια αντίδραση, μια πιο φιλόδοξη και ε, θαραλέα αντιμετώπιση ε, από αυτή την απάντηση που μας δίνει συνήθως η Κομισιόν ότι δηλαδή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ε, πράγμα που δεν είναι απόλυτα αληθές. Από τη στιγμή που στις διάφορες ε, εκθέσεις μας η Κομισιόν μπορεί να γνωρίζει τις προτάσεις βελτίωσης για τις πολιτικές εφαρμογές, έχω τα εξής ερωτήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη. Τα θέματα τα οποία τίθενται και που εμείς φωτίζουμε στην έκθεσή μας είναι πώς θα μπορέσουμε, μάλλον ποια μέτρα εσείς προβλέπετε ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις για τη μεταγραφή των ευρωπαϊκών νομοθεσιών στον δίκαιο των κρατών μελών. Είναι κάτι το οποίο λένε και ε, επιδεινώνεται, γιατί Όσο πιο αργά εφαρμόζονται οι νομοθεσίε, τόσο λιγότερο αποτελεσματικέ είναι. Πώ τότε μπορούμε να παίξουμε εμεί σωστά το ρόλο μα. Πώ επίση θα πρέπει να ενεργήσουμε ώστε να αιτιολογήσουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο η διαδικασία του 263 για τις εξηγήσει που υποχρεούνται να δίνουν τα κράτη-μέλη σε περίπτωση μη εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εν γέννη, πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση όσον αφορά τη μεταγραφή και μετά και την καλύτερη τη εκτέλεση τη νομοθεσία. Αυτό όσον αφορά την πρόληψη. Και επίση, πριν από 1,5 χρόνο, η Κομισιόν δημοσίευσε μία ανακοίνωση που λέει καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα. Όπου υπήρχε ένα πλάνο δράση ακριβώ για να καταφέρουμε να έχουμε περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Ποιον απολογισμό μπορείτε να κάνετε εσεί μετά από ένα χρόνο. Και έπειτα, όσον αφορά κυρώσει ή διορθώσει, αποκατάσταση, ε, υπάρχουν και τα εργαλεία του διαλόγου, για τα της τις συνεδριάσεις της επαφής ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Αυτά είναι χρήσιμα, γιατί έτσι καθίσατε η διαδικασία πιο διαφανής, αλλά και επειδή μπορεί να ε, έχουμε περισσότερα αποτελέσματα όσον αφορά την ταχύτερη μεταγραφή, αλλά και την ε, ε, καλύτερη εκτέλεση των νομοθεσιών. Και τέλος, ναι, όσον αφορά τις ε, διαδικασίες κατά παράβαση. Βλέπουμε, όπως έλεγα από την αρχή, ότι υπάρχει μια ε, σχετική ελαφρότητα ή ευαρέσκεια απέναντι στα κρατημέλη ε, χαλαρότητα. Εσείς από το Κοινοβούλιο έχετε μία πολιτική στήριξη. Ένα θεσμό που στηρίζει δηλαδή την Κομισιόν στο ρόλο της ε, ως θεματοφύλακα των συνθήκων, ως εγγυητή της σωστής εφαρμογής του δικαίου. Πώς να σας στηρίξουμε λοιπόν όσο περισσότερο μπορούμε να έχετε την ε, πολιτική νομιμότητα. Εντάξει, δεν χρειάζεστε απαραίτητα, αλλά ε, εμείς την ε, επικυρώνουμε ώστε να εγγυηθούμε στους πολίτες την καλύτερη και ορθότερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και τα δικαιώματά τους <clears throat> επίσης. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμανς, χαίρομαι που είστε μαζί μας γιατί πραγματικά μπορούμε να διεξάγουμε ένα σοβαρό διάλογο. Ε, θα θέσω δύο θέματα που έχουν σχέση με τις αναφορές, τις οποίες λαμβάνουμε, και θα επικεντρωθώ όμως στις ευρωεκλογές. Έχουμε πάρει αναφορές όπου οι πολίτες ε, σε διάφορες περιοχές και κάτοικοι διαφόρων περιοχών διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Οι, Ευρω... οι Βρετανοί ήθελαν να μπορούν να ψηφίσουν παρότι ζούσαν εκτός Βρετανίας. Σε άλλες περιοχές έχουμε α, κατοίκους οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν σε ευρωεκλογέ. Εγώ τώρα θα σας βάλω ένα άλλο ζήτημα που έχει σχέση με την επέκταση του σώματος το οποίο μπορεί να ψηφίσει. Δηλαδή, και έχει σχέση αυτό με την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Παλαιότερα όταν είχα ασχοληθεί πριν 20 χρόνια ως καθηγητής με το ζήτημα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, ε, είχα θέσει το ερώτημα αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε η Κομισιόν είτε άλλο κράτος μέλος, να ελέγξει υπό ποιους όρους ένα άλλο κράτος μέλος χορηγεί την υπηκότητά του Δηλαδή υπό ποιους όρους γίνεται κάποιος Έλληνας πολίτης. Αυτό το αποφασίζει μόνο η Ελλάδα, Φερρυπίν. Έχει δικαίωμα η Κομισιόν να θέσει ερωτήματα. Έχει δικαίωμα ένα άλλο κράτος μέλος να θέσει ερωτήματα. Και θα πείτε γιατί το λέω. Γιατί καθώς χορηγεί κανείς την υπηκότητα της Ελλάδος, ταυτόχρονα αποκτάει αυτός και την, την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Και έτσι λοιπόν ως Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να κινείται ελεύθερα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Το ερώτημα λοιπόν είναι, είναι δυνατόν και με ποιες διαδικασίες ένα κράτος μέλος να χορηγεί πλέον το δικαίωμα του πολίτη σε μετανάστες και με ποιους όρους, αλλάζοντας έτσι το εκλογικό σώμα. Παράδειγμα, στην Ελλάδα το εκλογικό μέτρο για να εκλέξει κάποιος ένα ευρωβουλευτή είναι περίπου 180 με 200.000 ψήφοι. Εάν ε, η κυβέρνηση δώσει το δικαίωμα ξαφνικά να γίνουν Έλληνες πολίτες 500.000 μετανάστες, αυτοί θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές και φυσικά να ψηφίσουν και έτσι μπορεί να εκλέξουν και δύο και τρεις ευρωβουλευτές. Ταυτόχρονα οι πολίτες αυτοί που θα είναι Έλληνες πολίτες είναι και Ευρωπαίοι πολίτες. Και άρα αποκτούν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και άρα έχουν και άλλα δικαιώματα κυκλοφορίας, εργασίας στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δικαίωμα η Κομισιόν να ελέγξει υπό ποιου όρου χορηγείται μαζικά πλέον η ηθαγένεια σε αυτό το κράτος. Και το λέω γιατί στην Ελλάδα σε ένα χρόνο έχουμε εκλογές η κυβέρνηση αρχίζει μια διαδικασία μαζική ελληνοποίησεων, χορήγησης της ε, ελληνικής ηθαγένειας σε πάρα πολλούς χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα. Σας λέω ότι το 2016 33.000 Αλβανοί έγιναν Έλληνες πολίτες. Ε, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση παραμονές εκλογών είναι λίγο προβληματική, διότι αλλάζει το εκλογικό σώμα και ξαφνικά 800.000 άνθρωποι μπορούν να ψηφίσουν. Και προφανώ θα ψηφίσουν το κόμμα το οποίο με γρήγορε διαδικασίε του δίνει την ελληνική ηθαγένεια. Και έτσι λοιπόν αυτό επηρεάζει και το εκλογικό σώμα, επηρεάζει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα μπαίνει το ερώτημα έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει αυτές τις διαδικασίες μια και αυτοί οι ίδιοι οι μετανάστες γίνονται ταυτόχρονα και European citizens και άρα έχουν και άλλα δικαιώματα. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο δεν ξέρω αν μπορείτε να μας απαντήσετε. I have spoken only minutes. I have counted... Μόνο τέσσερα λεπτά μίλησα. Μέτρησα πριν έναν σοσιαλιστή που μίλησε 5,5 λεπτά. Συνεχίζω λοιπόν στα αγγλικά. Τη εξίσου σημαντική που έχει σχέση με το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελεύθερη έκφραση αυτή τη στιγμή των Ευρωβουλευτών. Εμείς είμαστε στο ECR, είμαστε η τρίτη σε δύναμη πολιτική ομάδα και όμως στην Ελλάδα δεν μας αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε πάνελ, σε τηλεοράσεις, ε, με βάση τη δύναμη που έχουμε, ότι είμαστε η τρίτη πολιτική δύναμη. Αν θέλουν μας καλούν στην κρατική τηλεόραση, αν θέλουν μας καλούν στην τηλεόραση της Βουλής, αν δεν τους αρέσει αυτά που λέμε σε εκπομπές της τηλεόρασης της Βουλής, τότε κατεβάζουν και το βίντεο το οποίο έχουν αναρτήσει και το εξαφανίζουν και σε άλλα ιδιωτικά κανάλια δεν μας δίνουν καν τη δυνατότητα να εμφανιστούμε. Και μπαίνει ένα θέμα. Μιλούμε για δημοκρατία, μιλούμε για ελευθερία έκφρασης, έχουμε τέτοιες αναφορές. Εμείς ως υποψήφοι στο μέλλον αλλά και ως ευρωβουλευτές τι δικαιώματα θα έχουμε όταν μας φημώνουν, όταν δεν μας δίνουν το δικαίωμα να εμφανιστούμε, όταν δεν υπάρχει πλουραλισμός. Τα λέω αυτά λοιπόν, I'm going to finish in 20 seconds. Ε, τα λέω αυτά λοιπόν γιατί είναι πολύ σημαντικά. Βαδίζουμε σε ευρωεκλογέ και η τράπουλα είναι σημαδεμένη και δεν μας δίνουν την ευκαιρία να εκφραστούμε και δεν μας δίνουν την ευκαιρία να είμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τα opinion polls τα οποία υπάρχουν είναι στημένα. Δεν κάνουν καν ερώτηση για το κόμμα μας το οποίο είναι καινούργιο να δούμε τι ποσοστά θα πάρει. Ρωτούν οι άσχετα κόμματα τα οποία δεν εκπροσωπούνται ούτε στη Βουλή ούτε στην Ευρωβουλή. Είναι λοιπόν μια παράγκα ένα στήσιμο το οποίο είναι επικίνδυνο. Και εγώ οφείλω να το πω και σε εσά, μια και συζητούμε για τα δικαιώματα των πολιτών, τα οποία είναι συνυφασμένα και με το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε. Ευχαριστώ πολύ. You know, colleagues, there is a point in being... Η Πρόεδρος, υπάρχει κάποιο νόημα στο να λαμβάνει κανείς το λόγο και κάποια στιγμή να τον επιστρέφει, έτσι, το μικρόφωνο δηλαδή. Σύσταση λοιπόν, πάρτε τον λόγο και μετά να τον επιστρέψετε. Αυτό δείχνει και ευγένεια προς τους συναδέλφους σας. Ο κύριος Τερικάβρας. Θα είμαι σύντομος, ελπίζω. Τρία ζήτηματα. Πρώτο. Τονίζω αυτά που είπε προηγουμένως η συνάδελφός μου από σοσιαλιστές και δημοκράτες. Στην ανακοίνωσή σας για την βελτιωμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη βελτίωση της εφαρμογής της φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρετείται από το ρόλο της ως θεματοφύλακα των συνθήκων, αφήνοντας την εφαρμογή της συνθήκης στα εθνικά δικαστήρια. Αυτό φαίνεται, λέω. Θα ήθελα να μάθω τι ε, γνώμη έχετε. Διότι εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας με τις αρχές των κρατών μελών για έρευνες που έχουν σχετικά με την εφαρμογή και συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αλλά νομίζω παρόλα αυτά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει τον ισχυρό τη ρόλο και να λέει και τον τελευταίο λόγο. Αντιθέτω, εσείς εμφανίζεστε, αυτοεμφανίζεστε ως περιττή. Δεύτερο, τι γνώμη έχετε σχετικά με τη δυνατότητα μιας διαφορετικής ερμηνείας του άρθρου 51 του Χάρτου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε, μιλούμε για την ε, Βρετανική ε, υπόθεση. Και ένα τρίτο σε κάποια κοινοβουλευτική επιτροπή είπατε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είπατε επιλέξει μην περιμένετε και πάρα πολλά σχετικά με τη μεταρρύθμιση Τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Αυτά είναι τα λόγια σας. Εγώ κάπως ανησύχησα, διότι δεν θα ήθελα να είναι πολύ χαμηλέ οι προσδοκίε μας. Ξέρω ότι τώρα ε, προχωρούμε στις, στις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Τι νομίζετε να υπάρχει ανεξάρτητος φορέας για την καταγραφή των πρωτοβουλειών, ώστε να μην τις κρίνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως είναι καλύτερα. Γιατί όχι όμως, γιατί όχι. Γιατί ωραία είναι να έχετε εσείς ε, την κρίση, αλλά δεν είναι και τόσο αντικειμενικό. Και ακόμη και η δυνατότητα να φανείτε πιο ενεργή πιο δραστήριοι στην συνέχεια που δίνεται, στο follow-up, διότι γνωρίζουμε ότι είναι ένα από τα προβλήματα, από προβλήματα των ευρωπαϊκών Πρωτοβουλίων πολιτών, που λίγε ολοκληρώθηκαν και πολλοί ακόμα λιγότερε ολοκληρώθηκαν θετικά. Μπορούμε να λέμε εμεί ε, στου πολίτες μας, είμαστε μαζί σα και να προχωρήστε, κάντε κτλ. Αν όμω, βγαίνουν, μαζεύουν υπογραφέ και τελικώ δεν γίνεται τίποτα, αυτό μάλλον ε, του οδηγεί στην απογοήτευση και μειώνει τον ενθουσιασμό τους. Θα ήθελα δύο λόγια γι' αυτό. Ευχαριστώ που ήρθατε να μας δείτε. Ευχαριστώ τελικά μα, Εδώ ολοκληρώθηκε ο γύρος των συντονιστών. Τώρα μπορούν να λάβουν το λόγο άλλα μέλη, όμως χρονόμετρο. Ένα λεπτό ο καθένας. Ο κ. Μαρινόφ. Ευχαριστώ συναδέλφους ε, συντονιστές ε, που ελευθέρωσαν το χώρο ώστε να μπορέσουμε και εμείς να θέσουμε κάποια ερωτήματα που μας απασχολούν και θα το εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι είστε εδώ και θα σας ρωτήσω κάτι που είναι πολύ ε, πιο ευρύ από τη λειτουργία της Επιτροπής μας. Θέλω να σας ρωτήσω για τη χθεσινή ανακοίνωση ποιοτική αλλαγής στη σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ταμείων και του κράτους δικαίου. Όσο πιο σύντομα το πείτε, όσο περισσότερα πείτε, ε, τόσο καλύτερα. Γιατί η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει. Ε, κατηγορίες ε, πολιτικοποίησης λέγεται πως πρόκειται για μια συναισθηματική ε, ανακοίνωση ε, είναι δημοφιλής στους πολίτες ε, στο βορρά, στο νότο, στην Ανατολή και στη Δύση. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος. Είμαστε υπό παρατήρηση. Εξορισμού έχουμε προβλήματα με το κράτος δικαίου. Πώς λοιπόν θα συνδυάσετε αυτό το μηχανισμό με το νέο. Ειλικρινά, πιστεύω πως πρέπει να ξεφορτωθείτε τον παλαιό ανεπιτυχή μηχανισμό παρακολούθησης και να συνεχίσετε με το νέο. Δεν μπορούν να συνεπάρχουν λογικά, γιατί εξ ορισμού θεωρούμαστε ένοχοι. Πώς θα το ξεπεράσετε αυτό το πρόβλημα. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η κυρία Καμπεσόν Ρουίς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για τρία ζητήματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε τριμερή διάλογο σε πλαίσιο των διαπραγματεύσεων γιατί ο Ευρωπαϊκό Σήμα ε, αναπηρίες. Ε, εδώ σε αυτή την ε, επιτροπή μας ενδιαφέρουν πολύ το θέμα. Είναι πολλά, πολλές οι αναφορές που μας έρχονται από ανθρώπους με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες. Έχω σας ρωτήσω, αυτό το σήμα μπορεί να θεωρηθεί ως διάκριση κατά των ανθρώπων με αναπηρίες και το εξηγώ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε έναν κοινό ορισμό του τι είναι η αναπηρία, η ειδική ανάγκη. Ε, έχουμε διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με το κράτος μέλος. Ε, το, για τον καθορισμό του κατά πόσο κάποιο είναι ανάπηρο ή όχι. Και αυτό μπορεί να έχει συνέπειε οικονομικέ, αλλά εφόσον μιλάμε για ευρωπαϊκό, ε, ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρία, ώστε να μην έχει προβλήματα στην περίπτωση που θελήσει να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη, πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ένας άνθρωπος που θεωρείται ανάπηρο στην Ισπανία δεν θα έχει προβλήματα αν πάει α πούμε στη Ρουμανία εφόσον ε, τα κριτήρια ας πούμε είναι πιο αυστηρά ή διαφορετικά και δεν θα υποστεί διάκριση εναντίον του σε σχέση με κάποιο Ρουμάνο ε, πολίτη. Πώς θα κάνουμε έτσι ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους διακρίσεις. Το άλλο είναι η ψήφο. Ξέρουμε ότι στις ευρωπαϊκές εκλογές η Κομισιόν εργαζόταν για να μπορέσει να διευκολυνθεί η ψήφο για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, με αναπηρία ιδιαίτερα για την άρση των αρχιτεκτονικών ε, εμποδίων. Όμως, ε, θα πρέπει να δούμε όμως και πάλι εκεί δεν υπάρχει ομοιόμορφη νομοθεσία εξετάζεται το ίδιο πρόβλημα και στο πλαίσιο του ΟΗΕ και πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια ώστε τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τους αυτούς τους ανθρώπους και δεν ξέρω αν θα ήταν σωστό να πιέσουμε στις επόμενες ευρωεκλογέ να ε, ε, θεσπιστεί μια στρατηγία, στρατηγική ώστε οι άνθρωποι αυτοί με ειδικέ ανάγκες ή με αναπηρίες να μπορέσουν να ψηφίσουν ε, να υπάρξει μια εξατία ευαισθητοποίηση στα κράτη-μέλη ώστε να βελτιώσουν βελτιώσουν τις σχετικές τους και να μπορέσουν να ψηφίσουν οι περισσότεροι άνθρωποι που υποφέρουν από αναπηρίες, και, αν όχι και όλοι. Και τέλος, μεταφορές. Μεταφορές είναι πρόβλημα για τους ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες. Διαρκώς έχουμε αναφορές για αυτό το θέμα. Ξέρω πώς εργάζεστε για εθελοντικές ε, ε, ρυθμίσεις, όμως... Σε όλα τα κράτη-μέλη δεν γίνονται οι ίδιες, δεν ισχύουν οι ίδιες και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνο επιθελοντικής βάσης. Θέλω να γνωρίζω λοιπόν να σκοπεύετε να κάνετε κάτι γιατί και οι άνθρωποι με αναπηρία πρέπει να έχουν ας πούμε κάποιο συνοδό για να μπορέσουν να πετάξουν ένα απλό παράδειγμα. Πρέπει ε, οριστικώς να αρθούν τα εμπόδια και οι φραγμοί ώστε να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να μετακινούνται. Ευχαριστώ Σολεντάδ. Ο κύριος ε, Owens. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ήθελα να ρωτήσω κάτι και την πλατφόρμα online. Ε, υποτίθεται θα δούλευε ήδη από το τέλος του προηγούμενου μήνα. Έχει ανέβει, λειτουργεί, είναι, μπορούν να μπουν οι πολίτες, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν, να την διερευνήσουν και για κάτι πιο τεχνικό. Ξέρετε τι software έχει χρησιμοποιηθεί για την πλατφόρμα αυτή, είναι open source ή κάτι άλλο γιατί έχουμε συζητήσει κάποιες ομάδες το θέμα αυτό ε, του software open source ε, εδώ στην, ε, στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ξέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, χαίρομαι πολύ που είστε και πάλι εδώ. Συναντηθήκαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για τα θέματα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων Ξέρετε ότι έχουμε ένα ψήφισμα σχετικά από την Επιτροπή μας και πάλι σας ευχαριστώ για, την, για το χρόνο που μας διαθέσατε και για την επιθυμία να συνεχίσετε τον διάλογο αυτό. Έχω δύο σύντομα ερωτήματα και πολύ συγκεκριμένα και εύκολα. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα εσωτερικό στην Επιτροπή μας την προηγούμενη εβδομάδα Είχαμε αιτούντε από την Λετωνία και την Εστονία εδώ και το ερώτημα ήταν τον, το, δικαίωμα πολι, μη πολιτών στην ε, Εστονία και την Λετωνία στις ευρωεκλογέ. Η θέση σας ποια είναι για αυτούς τους ανθρώπου. Ξέρω ότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, πολύ περίπλοκο. Και δεύτερο ερώτημα, το θέμα του Brexit. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές σχετικές για τα, με τα δικαιώματα των ε, Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στην ε, ε, Μεγάλη Βρετανία και Βρετανών υπηκών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και μια πολύ ισχυρή αντιπροσωπεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθηγητές της οποίας προείδρευα εγώ και μας είχαν ζητήσει τότε να δούμε πώς γίνεται να τους βοηθήσουμε εμείς εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί για το θέμα του τι θα γίνει με την έξοδο της, Ευρωπαϊκής, της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους είπα ότι το θέμα είναι στα χέρια σας. Εσείς πρέπει ίσως να κάνετε ένα δεύτερο δημοψήφισμα για το έγγραφο της συνθήκης αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική σας άποψη ποια είναι. Έχετε κάποιες τέτοιες σχέσεις για ένα πιθανό ίσως ε, δεύτερο νέο δημοψήφισμα. Και ίσως να είμαι και ο μόνος εδώ στο Κοινοβούλιο που, να, που λέω ότι το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει με τον Brexit. Ίσως να είναι ακόμα ανοιχτό και να μπορούμε με κάποιο τρόπο να το λύσουμε. Ε, καλό είναι να υπάρχει και κάποιος αισιόδοξο εδώ ανάμεσά μας. Well, μετά από την στήριξη του, της ψήφου των ε, πολιτών για το θέμα του Brexit στον Ηνωμένο Βασίλειο, που την χάνει όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη, δύο ερωτήματα έχω. Καταρχάς, ακούσαμε τα σχόλια για το θεμελιώδες θέμα των, ε, του δικαιώματος του εκλέγην και εκλέγεστε και για το Brexit, για με τον Brexit, πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία θα δούμε ότι υπάρχει όντως, ε, θα υπάρξουν ίσως πολίτες που δεν θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε εσείς ως Επίτροπος υπεύθυνο για τα δικαιώματα των πολιτών, τι πιστεύετε για την πολιτική του συμμετοχή σε αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία αποχώρησης θα καλύπτει και πολιτικά δικαιώματα και οικονομικά δικαιώματα των πολιτών και στις δύο πλευρές του καναλιού. Και επίσης έχω να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπε η Βερζινή για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει όρεξη να προωθήσει κάποιες μακροχρόνιες ε, διαδικασίες υπερβάση που υπάρχουν. Ε, έχουμε κάποιες ε, διαδικασίες που κρατούν δεκαετίες. Ε, πολίτες προσπαθούν να βρουν το δίκαιο τους εδώ και δεκαετίες. Ας πούμε έχουμε έτης, αναφορά από την Ιταλία. Έχουν κερδίσει έξι υποθέσεις παραβίαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και παρόλα αυτά κάθε φορά η Ιταλική κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι θα υπάρξει διακριτική μεταχείριση στο, στους ακαδημαϊκούς χώρους για τους αλλοδαπούς καθηγητές. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε, λέκτορες. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα θέματα αυτά που πραγματικά υπονομεύουν την ε, αξιοπιστία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μητροβάνοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμανς, Είστε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εμείς είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ξέρετε ότι παρόμοια ερωτήματα λαμβάνουμε και εμείς. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά τόσο δυνατά στα οικονομικά θέματα, αλλά είναι τόσο δύναμη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί να εξασφαλίσει ε, ισότητα των ε, δικαιωμάτων των πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λάβει πολλές αναφορές για, την, για τα δικαιώματα ψήφου στην ε, Λετωνία και την ε, Εστονία από μη πολίτες. Και μιλούμε και για το θέμα της ε, έλλειψης υπηκότητας. Αυτή την άνοιξη θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε ε, αναφορές πάλι από την ε, Λετωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για, την, ε, για το δικαίωμα ε, εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα. Ίσως λοιπόν η Κομισιόν πρέπει να δράσει λίγο πιο αποτελεσματικά και πιο ενεργητικά για να δημιουργήσει έναν ε, διάλογο με τα κράτη αυτά για τα θέματα της επικότητας, της ηθαγένειας, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της, εκπαίδευσης, της δυνατότητας εκπαίδευσης του στη μητρική τους γλώσσα. Ευχαριστώ κύριε Βίλαντ. Καλώς ήρθατε. Θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που βγήκα για λίγα λεπτά. Έχω νέα. Ε, με υπεγράφησαν, αλλά δεν εξηγεί τι ακριβώς ο κύριος Βίλαντ. Έγινε υπογραφή κύριε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Έχουμε αποφασίσει ορισμένα πράγματα και θέλω να έρθω να τα συζητήσω μαζί σας. Ακούω από δικαστές και φτάνουν και στην Επιτροπή Αναφορών. Ότι δηλαδή είναι ένα είδος αναθεωρητικής αρχής η Επιτροπή Αναφορών. Όμως πολλά πράγματα φτάνουν εδώ διότι δεν ικανοποιούνται και από την ομολογία οι πολίτες. Ακούω από το δικαστήριο παράπονα ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μεταφράσεων των ε, κειμένων που ε, χρησιμοποιούν ως βάση και των αποφάσεων και που επεξεργάζονται γενικά. Δεύτερο, ακούω για διαφορετικές πρακτικές στις χώρες μέλη σχετικά με την επίλυση διαφορών. για τη συνεργασία των τμήματων. Τρίτο, βεβαίως τώρα σας θέτω ε, ζητήματα ε, λεπτομεριών από μεμονωμένες αναφορές. Αλλά παίρνω μια αναφορά μεμονωμένα όπου δεν ε, την βρήκα τη λύση που δόθηκε ικανοποιητική. Έχουμε την περίφημη δροσόφυλλα μελανογκάστερ, εκείνη την μιγούλα που ζει μία μόνο ημέρα και όπου αποστολές τέτοιων εντόμων τα σταμάτησαν στα αεροδρόμια, τι αποστολές τα σταμάτησαν στα αεροδρόμια για να τις κριστάσουν οι κτηνίατροι. Βεβαίω, μια τέτοια μίγα ζει μονάχα μία μέρα, το λέει και το όνομά της στα, στα γερμανικά τουλάχιστον, μίγα τη μια ημέρα. Και έτσι φτάσανε στα επιστημονικά εργαστήρια τα δείγματα αυτά νεκρά. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να σας οδηγήσει στην αναθεώρηση όλων των βασικών κειμένων, όμως δεν έχει δοθεί και καμία λύση Πρόκειται για την αναφορά 1358 του 2011. Είναι μια αναφορά την υπογράφουν πολλοί επιστήμονες μεταξύ αυτών και βραβευμένοι με Νόμπελ και χρειάζεται να δοθεί κάποια κίνηση εκεί. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταμάτησε συνολικά ορισμένες διαδικασίες για παραβιάσεις των συνθήκων. Εάν κλείνει κάποια πράγματα. Για πολιτικού λόγου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι θεωρεί ότι η περαιτέρω διαδικασία δεν είναι σκόπιμη. Και πάλι, από την άλλη μεριά, εάν πάλι για πολιτικού λόγου θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν είναι σκόπιμο να κάνει κάτι. Μπορεί βέβαια τέλο πάντων να καταλήξει κανεί σε μια τέτοια άποψη. Έχω ακούσει όμω από εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου λένε ότι ναι, δεν είναι ακριβώ παραβίαση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Αυτά ήταν κάποιες λύσεις που, δώσανε, που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν ικανοποιούν τελικώς κανέναν. Θα πρέπει η θεμελίωση, η τεκμηρίωση να είναι πολύ πιο ισχυρή και ξεκάθαρη. Μάλιστα, σας ευχαριστώ όλους και όλου. Κύριε ε, Αντιπρόεδρε, δικό σα το δύσκολο καθήκον να δώσετε όσε περισσότερε απαντήσει μπορείτε. Ίσως μπορούμε να μείνουμε και λίγα λεπτά παραπάνω. υπηρετώ, εξυπηρετώ αν θέλετε πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ποτέ, και έρχομαι δηλαδή σε επαφή μαζί τους, ποτέ δεν μου θέτουν τόσο ευρύ φάσμα ερωτήσεων όσο η δική σας. Σαφώς καταθέτεται σήμερα στη συζήτηση πολλά από τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες στις αναφορές τους. Θα προσπαθήσω να δικαιώσω, τέλο πάντων να δώσω απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο ορισμένες δεν θα μπορέσω να τις απαντήσω ευθέως και αν μου επιτρέπετε θα σας τις απαντήσω γραπτός. Για το θέμα των ταχύτερων απαντήσεων στις αναφορές. Νομίζω ότι συνολικά έχουμε βελτιωθεί τα τελευταία λίγα χρόνια. Τα πράγματα κινούνται ταχύτερα από ότι ε, στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά θα επανεξετάσω το θέμα του πότε συμπεραίνουμε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι. Να δω αν μπορούμε εκεί να επιταχύνουμε. Να μπορούμε δηλαδή γρήγορα να απαντήσουμε στην περίπτωση αυτή. Μου θυμίζει κάτι το οποίο με απασχολεί και καθημερινά στο γραφείο μου λαμβάνω έναν απίστευτο αριθμό προσκλήσεων ε, να προσέλθω σε γεύματα, δείπνα, ε, διαλέξεις, ομιλίες και έχουμε μια πολύ ε, λεπτομερή διαδικασία ελέγχων, τη λέμε Green Fish Process, Είναι, υπάρχουν δηλαδή πολλές λεπτομέρειες που ρυθμίζουν και πριν να μπορέσω να απαντήσω, λέω στους ε, συνεργάτες μου, κοιτάξτε πρώτα το ημερολόγιο, την ατζέντα, εάν μπορώ να πάω ή όχι. Και επειδή ακριβώς ελεγχόμεθα και αντικειμενικά, αντικειμενικά ε, δικαιολογημένος έλεγχος, δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη. Και καμιά φορά προσπαθώντας κανείς να αποφύγει λάθη, ε, καθυστερεί. Δηλαδή αυτό, αυτό αποβαίνει σε κόστος της ταχύτητας της αντίδρασης. Εάν λοιπόν δεν είμαστε αρμόδιοι και το γνωρίζουμε αυτό εξ αρχής, μπορούμε ίσως να απαντήσουμε ταχύτερα. Θα επανέλθω σε αυτό, εάν μπορούμε πράγματι να κάνουμε κάτι εκεί. Πολλοί, πολλοί εξημών έθεσαν το θέμα των παραβιάσεων, των διαδικασιών παραβιάσεων. Νομίζω οι μισοί από σας έθεσαν το θέμα αυτό. Διερωτώ με λοιπόν, εάν υπάρχει κάπως ευρύτερο πρόβλημα, αφού τόσο πολλοί εξημών το θέσατε. Η πρόταση που θα κάνω εγώ για το θέμα αυτό είναι να μου επιτρέψετε να το αναλύσω λίγο περισσότερο. Ε, το πρώτο μου ένστικτο είναι να πω όχι, ε, διότι έχουμε ένα τεράστιο αριθμό διαδικασιών παραβιάσεων. Ας το ξαναδώ και ας επανέλθουμε, να σας δώσω μια συνολική επισκόπηση, να ενημερωθώ και από τις υπηρεσίες μου, εάν υπάρχει ίσως κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε περισσότερο. Δεν έχω καμία ένδειξη, αλλά και μόνο από το γεγονό ότι τόσο πολύ θέσατε το θέμα ε, με κάνει να πω μια στιγμή, Α το ξαναδούμε, α το δούμε πιο κοντά. Και μπορούμε ίσω να επανέλθουμε όταν ε, θα το έχουμε δει. Διότι θα συμφωνήσω με την άποψη που εφράσατε ορισμένη ότι η αξιοπιστία των θεσμικών μας οργάνων εξαρτάται μεταξύ άλλων και από την δίκαιη και πλήρη εφαρμογή, η ανταπόκριση τέλο πάντων στις ευθύνες μας. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε το στοιχείο της διάκρισης, αν θα θελήσει κανείς να προωθήσει μια διαδικασία παραβίασης ή όχι. Όμως διακριτική αυτή ευχαίρεια θα πρέπει να είναι θεμελιωμένη νομικά. Διότι εφόσον υπάρχει παραβίαση δικαίου, καλείται το θεσμικό όργανο να την αντιμετωπίσει και δεν μπορεί να πολιτικοποιηθεί το θέμα αυτό. Να, α, πολύ δύσκολο θέμα, α, πολύ πολιτικό αυτό, α το αφήσουμε στην άκρη θέματα όπως η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που θέσατε πριν. Πρόκειται για αποφάσεις σοβαρότατες, αλλά δεν θα αποφύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τις αποφάσεις αυτές. Άλλωστε βρισκόμαστε εν μέση διαδικασία εξέτασης των ε, αποφάσεων αυτών. Και για άλλα θέματα, ιδίως όσα έχουν ε, με σχέση με την ε, δημόσια υγεία. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εφόσον θίγονται θέματα περιβάλλοντος. Η έκθεση που λάβαμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σχετικά με το πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Και μιλούμε για θανάτους, δεν μιλούμε απλώς για βλάβη της υγείας. Και εάν έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαιτεί από τις χώρες μέλη να διατηρούν ένα κάποιο επίπεδο ε, ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ούτω ή άλλω αυτέ το αποφάσισαν. Οι χώρε το αποφάσισαν. Δεν ε, είμαστε δικτάτορε που σα επιβάλλουμε κάτι. Μαζί σα, δηλαδή με το Συμβούλιο Υπουργών, αυτό συναποφάσισε. Ενέκρινε την νομοθεσία αυτή. Και επομένω, σωστό είναι να του θεωρήσουμε υπόλογου. Σα ευχαριστώ για την πρόταση λοιπόν. Ε, θα εγκύψω και θα δω αν μπορώ να σας δώσω κάτι να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά τα γεγονότα θα μιλήσουν μόνα τους και θα δούμε όταν θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Εξάλλου, έχουμε ήδη κάτι το οποίο λειτουργεί καλύτερα και από ό,τι εγώ νόμιζα αρχικά. Δηλαδή η πλατφόρμα Refit που νομίζω ότι είναι και κάπως μοναδική. Οι χώρε μπέλη δεν έχουν τέτοια πράγματα. Όταν εξετάζουμε δηλαδή την υφιστάμενη νομοθεσία και, κοιτούμε εάν πραγματικά τα αποκρίνεται στους στόχους, στις ανάγκες, θα έλεγα ότι το δίκτυο αναφορών μπορεί πράγματι να δώσει κάποια εναύσματα και για την ε, διαδικασία REFIT. Πολύ καλό θα ήταν λοιπόν να συναποτελέσει μέρος ε, του διαλόγου μας. Η πλατφόρμα Refit, ε, σε αυτήν συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη από όλες τις χώρες μέλη. Είναι δηλαδή ένα είδος ε, συμπυκνωμένης μορφής αναφορών, ειδικότερα βέβαια για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και για πτυχές ευρωπαϊκής νομοθεσίας που δεν αποδίδουν στην πράξη. Τώρα η καθυστερημένη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαδικασιών για παραβίαση εφόσον αυτό χρειαστεί. Και θα πρέπει να δούμε, να σημειώσουμε ότι και η περιπλοκότητα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας έχει αυξηθεί σημαντικά. Κάτι το οποίο καθιστά και την μεταφορά στα εθνικά δίκαια ακόμα πιο περίπλοκη χωρίς να αποκλείω όμως ότι δεν είναι μόνο η περιπλοκότητα που παίζει κάποιο ρόλο, αλλά ενδεχομένω και κάποια ζητήματα πολιτικών σκοπιμοτήτων που δεν μπορώ να αποκλείσω. Άρα χρειάζεται στενή και συστηματική παρακολούθηση και μεταξύ άλλων και του γεγονότος ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται στο Εθνικό Δίκαιο οι οδηγίες θα πρέπει να ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ελέγχεται και από το Κοινοβούλιο. Αν θέλουμε λοιπόν να γίνει ε, ένα είδος καταγραφής αυτών, νομίζω ότι μπορεί να γίνει με τον τρόπο που εξήγησα. Τώρα, σχετικά με τις εκλογές και την χορήγηση της θαγένειας, ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα. Περίπλοκο διότι και η απόφαση σχετικά με το ποιος επιτρέπεται να ψηφίσει, να συμμετάσχει στις εκλογές και ποιος λαμβάνει την εθνική ηθαγένεια, ως γνωρίζετε είναι εθνική αρμοδιότητα. Έχουμε, έχουμε ευρωπαϊκά πρότυπα βεβαίως και βρισκόμαστε και μέσα σε μια συζήτηση για αυτό το λεγόμενο passport scheme στη Μάλτα. Έχουμε κάποιες απαιτήσει, όταν δηλαδή δώσετε ηθαγένεια σε κάποιον πρέπει να έχει κάποια προφανή διασύνδεση με τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό απαιτείται. Τώρα απλά μαζική χορήγηση ηθαγένειας φαίνεται όντω να αντιβαίνει σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Το διατυπώνω πολύ προσεκτικά. Ωστόσο, το δικαίωμα χορήγηση ηθαγένεια υπό ορισμένε συνθήκες, υπό ορισμένου όρου, είναι εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα των χωρών μελών. Έχουν όμως την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι το γεγονό ότι χορηγούν το δικαίωμα αυτό λαμβάνει υπόψη και τα συμφέροντα άλλων χωρών μελών, των άλλων χωρών μελών. Αυτά είναι ε, τα στάνταρ που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και φοβούμαι ότι δεν μπορώ να απαντήσω ευρύτερα από αυτό. Κύριε Μαριά, επίσης στο ίδιο πλαίσιο μιλήσατε για residency και citizenship, διαμονή και ηθαγένεια. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών και οι διαμένοντες στις χώρες ενώ μέχρι τώρα ήταν μόνο στη χώρα από την οποία κατάγεσαι. Θα μπορείς να ε, βάζεις υπογραφή και για χώρα στην οποία διαμένεις. Δεν γνωρίζω τους κανόνες των πολιτικών συζητήσεων στην ελληνική ε, τηλεόραση. Ομολογώ δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω εάν ε, υπάρχει κάποιος αποκλεισμός από την ε, ελευθερία των μέσων ειδικά σήμερα. Πάντως ε, η ελευθερία των μέσων είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ανησυχεί. Εάν δεν γίνεται σεβαστός ο ανεξάρτητος ρόλος των μέσων σαν ένα απαραίτητο θεσμικό εργαλείο της δημοκρατίας. Δυστυχώς αυτό είναι μια τάση την οποία βλέπουμε και βεβαίως όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ένα αριθμό χωρών μελών, αλλά και έξω από τις χώρες μέλη αυτές. Και οι πολιτικοί φέρουν τεράστια ευθύνη όταν από τη μια μεριά λέμε fake news ή διεφθαρμένα τα μέσα κλπ. Με τον τρόπο αυτό ωστόσο υπονομεύουμε έναν από τους βασικούς θεσμούς της δημοκρατικής κοινωνίας. Χρειάζεται λοιπόν πράγματι σεβασμός της ανεξαρτησίας των μέσων, γενικά το λεφτό, όχι μόνο ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, και την εφαρμογή την αφήνουμε στις χώρες μέλη. Το είπα αυτό σχετικά, μίλησα δηλαδή σχετικά γι' αυτό ήδη, άλλωστε θα επανέλθουμε σε αυτό, κάνουμε μια εσωτερική έρευνα για το άρθρο 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουμε μέτρα για τις παραβιάσεις και εάν αν παραβιαστούν τα άρθρα του χάρτη, όμω οι αρμοδιότητε μα δεν προκύπτουν από το χάρτη. Οι αρμοδιότητε μα προκύπτουν από τη συνθήκη και στην βάση αυτών ερμηνεύουμε και τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αν θέλουμε τώρα να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή του άρθρου 51, για αυτό ωστόσο θα χρειαστεί τροποποίηση τη συνθήκη. Χωρί τροποποίηση τη συνθήκη, αναθεώρηση τη βλέπετε, δεν μπορεί να γίνει. Υποστηρίζουμε τις ε, ε, οργανώσεις πολιτών και ούτω καθεξής. Γνωρίζουμε ποιες είναι και οι προσδοκίες των πολιτών στον τομέα αυτό. Δεν μπορούμε όμως να υπερβούμε τα όρια των αρμοδιοτήτων που μας επιβάλλει η συνθήκη. Για τον ανεξάρτητο φορέα για την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, να το πω ως εξής. Εάν Αυτό το συζητούσα πριν μαζί σας. Δεν είπα μην περιμένετε πολλά από τις αλλαγές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Είπα μην την, παρα, μην την πλασάρετε υπερβολικά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δεν αποτελεί εναλλακτική λύση σε δημοψήφισμα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί μια δυνατότητα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτε να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να νομοθετήσει σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Δεν του δίνει το δικαίωμα να ανακατευτούν στην νομοθέτηση. Αν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μα το ζητήσουν, βεβαίω αυξάνει το αίσθημα ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αναλάβει πρωτοβουλία στο συγκεκριμένο τομέα. Και όπω έχουμε κάνει. Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία πολιτών δεν έχει φτάσει ακόμα, δεν έχει εξαντλήσει το δυναμικό της. Μένει ακόμα δυναμικό. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες πολιτών που οδήγησαν σε κάποιο αποτέλεσμα οδήγησαν τελικώ στην λήψη μέτρων από εμάς ορισμένες φωνές νομοθετικών, όπως για την οδηγία περί πόσιμου νερού, ή και με παθητικό τρόπο. Και οι πρόσφατες αποφάσεις για την κατάργηση ορισμένων ζυζανιοκτώνων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην βιοπικιλία προκλήθηκαν, οι αποφάσεις αυτές, από μια πρωτοβουλία πολιτών. Νομίζω πάντως ότι στο σελίδα λειτουργεί, αν και δεν έχω σχετική πληροφόρηση. Αν όχι, τότε θα σας το γνωρίσω αμέσως. Τώρα για το λογισμικό ανοιχτή πηγής δεν ξέρω. Θα μάθω και θα σας πω. Ταμεία και κράτος δικαίου. Αυτά έχουν σχέση με το δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως η συνδρομή στις χώρες μέλη για να φτάσουν στο αναγκαίο επίπεδο προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων οι διαδικασίε που έχουμε με Βουλγαρία και Ρουμανία είναι διότι όταν οι χώρες μέλη αυτές εντάχθηκαν δεν είχαν φτάσει ακόμη στο επίπεδο του αγώνα κατά της διαφθοράς και στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που θα θέλαμε. Έχουμε ωστόσο κάνει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια και με σημαντική υποστήριξη μεγάλων τμήματων του πληθυσμού των χωρών αυτών. Ακούω, βλέπω μάλλον γκρινιάρικες κυβερνήσεις, αλλά ενθουσιώδεις πολίτες. Καλύτερα μου αρέσει έτσι πάντως παρά ανάποδα. Πάντως, τα δύο, οι δύο αυτοί μηχανισμοί μπορούν να ζουν και να συνεργάζονται. Διότι το στοιχείο του κράτους δικαίου στο δημοσιονομικό κανονισμό σημαίνει παράλληλα δηλαδή με το δημοσιονομικό Οργανισμό, σημαίνει ότι δεν μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται ορθά, εάν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ανεξάρτητη δικαιοσύνη που θα το ελέγξει. Μιλούμε δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων. Και για να είναι απόλυτα σαφές. Εάν υπάρχει τέτοια διαδικασία, δεν απαλλάσσει αυτό η χώρα μέλος από την ευθύνη να χρηματοδοτεί έργα. Δηλαδή οι δικαιούχοι των χρημάτων δεν θα ε, υποστούν ζημία. Διότι θα παραμείνουν υπεύθυνε υπόλογε οι κυβερνήσει για να χρηματοδοτήσουν τα έργα. Αυτό θα είναι ο μηχανισμό. Για να δούμε πώ ακριβώ δαπανώνται τα χρήματα, τα ευρωπαϊκά χρήματα. Και αυτό δεν αναφέρεται μοναχά στο Ταμείο Συνοχής, αλλά πρόκειται για όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τώρα ζητήματα αναπηριών. Έχουμε δουλειά να κάνουμε πριν από τι επόμενε ευρωεκλογέ και εγώ θα είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο να μπορέσουμε να πούμε αληθώ όμω, ότι οι ανάπηροι άνθρωποι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν απρόσκοπτα στι επόμενε ευρωεκλογέ. Θα ήθελα να υπάρχει ήδη η ε, οδηγία ισότιμη μεταχείριση να έχουμε δηλαδή πλήρη πρόσβαση σε δημόσια κτίρια και ούτω καθεξής. Πάντως ενημερωνόμουν μόλις για τον τριμερή διάλογο, θα δω πώς μπορώ να βοηθήσω τους ε, συναδέλφους μου επιτρόπους για να σας βοηθήσουν και εσάς, θα τους μιλήσω και έχουμε βέβαια ακόμα σημαντικές προκλήσεις ό,τι αφορά την πρόσβαση σε δημόσιες ε, συγκοινωνίες, ιδίως ε, στις αεροπορικές και ούτω καθεξής και Νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε επιτύχει περισσότερα αν είχαμε ασκήσει μεγαλύτερη πίεση. Πάντως ευχαρίστω να συνεχίσω τον διάλογο για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Για τα δικαιώματα ψήφου σε Εστονία και Λετωνία. Μακρότατη, μακρότατο ιστορικό με το ζήτημα αυτό, έχοντας εργαστεί και στον ΟΑΣΕ στο παρελθόν, στα μέσα της δεκαετίας του 90 για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι δίκαιο, μπορώ να πω δηλαδή, ότι σε σύγκριση της κατάστασης της τότε με την τώρα έχει πράγματι γίνει ευκολότερο, πολύ ευκολότερο για μη υπηκόους να λάβουν την υπηκότητα και σε μεγάλο βαθμό νομίζω είναι και συνειδητή επιλογή τους να μην γίνουν τελικά επίκοοι. Και αν βεβαίως λάβουν την απόφαση αυτή συνειδητά, αυτό βεβαίως έχει συνέπειες στα εκλογικά τους δικαιώματα και σε άλλα δικαιώματα. Και γνωρίζω ότι στο παρελθόν ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κανείς πολίτης της Λετωνίας ή της Εστονίας λόγω των γλωσσικών απαιτήσεων, εξετάσεων, αλλά δεν συμβαίνουν τώρα πλέον. Πάντως όχι στον ίδιο βαθμό και ιδίω για τους νεότερους, οι οποίοι ε, είναι απολύτως Ε, Εκτός πλέον και αν είναι απολύτως αποκεκλεισμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία που κανείς δεν το θέλει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει πάντοτε να προσέχουμε ιδιαίτερα τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ακόμα και αν δεν είναι πολίτες μιας συγκεκριμένη χώρας ή ακόμα καλύτερα αν είναι απάτριδες, γιατί ορισμένοι από αυτούς δεν είναι ούτε των ε, δύο αυτών βαλτικών χωρών, ούτε της Ρωσίας. Χρειάζεται και θα χρειάζεται πάντοτε προσοχή και διάλογο με τι κυβερνήσει των δύο αυτών χωρών. Δεν μπορώ όμω να ασκήσω κάποια βαριά κριτική για την κατάσταση αυτή, διότι έχουν προσφέρει καλύτερη πρόσβαση τώρα. Στην Ιθαγένεια πάντοτε υπάρχουν θέματα εκπαίδευση στην γλώσσα των μειονοτήτων κλπ. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα αυτά πάντοτε. Αλλά μέχρι τώρα και με τρόπο επικοδομητικό οι δύο αυτέ χώρε μέλη μπόρεσαν να εξεύρουν διεξόδου. Αν υπάρχουν άλλα θέματα, ευχαρίστω θα θα ακούσω, θα ακούσω και αυτούς και εσάς, αλλά εύχομαι πράγματι τα δικαιώματα, μάλλον θα ευχόμουν τα δικαιώματα των Ρώσων πολιτών να ήταν το ίδιο καλά εγγυημένα όπως είναι στην Εστονία και στην Λετωνία. Γιατί πολλοί μη ηθαγενείς Εστονίας και Λετωνίας έχουν καλύτερα προστατευόμενα δικαιώματα από τους Ρώσους πολίτες για το Brexit, άμεση δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο, κάποια υψηλότερη αξία ενός δημοψηφίσματος από ότι της αντιπροσωπητής δημοκρατίας. Δεν κατανοώ γιατί άραγε το δημοψήφισμα να έχει μεγαλύτερη πολιτική ή ηθική βαρύτητα από την ψήφο στις εκλογές. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι το Βρετανικό Δημοψήφισμα για το Brexit δείχνει ότι καμιά φορά ένα ερώτημα που φαίνεται απλό κρύβει από πίσω μια περιπλοκότητα που δεν μπορούν πραγματικά να συλλάβουν οι άνθρωποι τη στιγμή που πάνε να δώσουν την απάντηση σε μια ερώτηση. Δίνουν μια απάντηση και μετά προκύπτει ότι η απάντηση που έδωσαν χωρίς να έχουν πλήρη, πληρέστατη ενημέρωση τότε κοίταξτε, διαρωτώ με ποια είναι η υψηλότερη μορφή δημοκρατία, αλλά μην το συζητήσουμε αυτό σήμερα. Εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται να κάνω τώρα εικασίε για επανάληψη δημοψήφισματος κλπ. Δεν είναι δικό μου ρόλο. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα σα τα είπα. Νομίζω ότι απάντησα και στις περισσότερες ερωτήσεις και τις δικέ σας και τις δικές σας. Για την τροσόφυλλα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Να επανέλθω γραπτός. Τα θυμάμαι από το γυμνάσιο. Φαίνεται σαν ένας αιώνα πριν, όπου στην βιολογία μας είχαν πει ε, για αυτά τα ζωήφια. Και απάντησα και για την πολιτική τεκμηρίωση των διαδικασιών παραβίασης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία αυτή η ανταλλαγής απόψεων και σας εύχομαι καλή ε, επιτυχία στις συνεχιζόμενες προσπάθειές σας και εμείς θα σας υποστηρίξουμε όσο μπορούμε. Το έγγραφο με τα συμπεράσματα της σημερινής συζήτηση ε, θα τα στείλουμε στους συντονιστές αύριο και στις 15 Μαΐου και 16 Μαΐου θα φτάσουμε στο τελικό κείμενο για να είμαστε και αποτελεσματικές και αποτελεσματικοί. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.